Αγαπητή Πρόεδρε, κυρία Κώστα, κυρία Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη του, είστε αυτοί που διαμορφώνετε τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν σας παρουσιάσω το δικό μου όραμα για αυτό το χαρτοφυλάκιο, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το λόγο που είμαι ευτυχής να βρίσκομαι εδώ απόψε. Το να είναι κανείς επίτροπος σημαίνει να είναι στρατευμένος Ευρωπαίος. Το να είναι κανείς επίτροπος σημαίνει να εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και κανένα άλλο συμφέρον. Το να είναι κανείς επίτροπο σημαίνει να υπηρετεί τον Ευρωπαίο πολίτη δεν μπορώ να σκεφτώ μεγαλύτερη τιμή, επομένως από το να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Γνωρίζετε και εσείς, γνωρίζω και εγώ, ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουγγαρίας ε, δήλθαν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Διαφωνήσαμε για συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα και εκφράσαμε τις αντιθέσεις μας ε, με έντονο τρόπο, με ηχηρό τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως, μια από τις μεγάλες αρετές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι μας δίνει το χώρο να ε, αντιπαραβάλλουμε τις διαφορές μας ε, και να λύσουμε τις διαφωνίες μας, αλλά με τρόπο ανοιχτό, δημοκρατικό και ειρηνικό να βρούμε μια λύση ε, στις διαφωνίες μας, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, μας κάνει πιο δυνατούς και σαν χώρες μεμονωμένα, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Εν τέλει, μας ενώνουν οι ίδιες ευρωπαϊκές αξίες. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για αξίες ε, στις οποίες είμαι βαθύτατα και προσωπικά δεσμευμένος. Απόψε θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το όραμα που έχω για την παιδεία, τον πολιτισμό, την νεολαία και την ηθαγένεια. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το έργο το οποίο πρέπει από κοινού να φέρουμε σε πέρας. Αν διαβάσετε ορισμένες από τις εφημερίδες μας, ίσως αποκομίσετε την εντύπωση ότι το λόγο χαρτοφυλάκιο δεν είναι και το πλέον επίγον. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ. Διότι ποια πρόκληση είναι πιο επίγουσα από το μέλλον της νεολαίας μας. Ποιο πρόβλημα είναι πιο ανησυχητικό από την ανεργία των νέων που παραμένει πάνω από το 50% σε ορισμένες χώρες. Ποιο καθήκον είναι πιο σημαντικό και πιο απαραίτητο από το να δώσουμε στις μελλοντικέ γενιές την καλύτερη δυνατή εκκίνηση ε, στη ζωή τους και τι μπορεί να είναι πιο πολύτιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την παιδεία, τον πολιτισμό της και την αίσθηση της ταυτότητας. Ποιοι τομείς πρέπει να τύχουν προστασίας ε, περισσότερο από τις πολιτισμικές διουρικές βιομηχανίες. Τι είναι η Ευρώπη αν δεν είναι κοινή κληρονομιά, μια κοινότητα κοινών αξιών. Αξιότιμοι βουλευτές, πιστεύω ότι το χαρτοφυλάκιό μας ε, είναι όσο ζωτικό όσο οποιοδήποτε άλλο. Αν θέλουμε να επανοικοδομήσουμε μια δίκαιη βιώσιμη οικονομία πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση, με την παιδεία. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους μας για έναν πολυπολιτισμικό και ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Αν θέλουμε οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί μας να βρουν νέο ακροατήριο ε, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να του δώσουμε τα εργαλεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να ανθίσουν στην ψηφιακή εποχή. Όλοι ε, θεωρούμε ότι η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η συμμετοχή στα κοινά είναι μέσω να απελευθερώσουμε το δυναμικό μας ως ανθρώπινα όντα. Δεν είμαστε οικονομικοί πόροι, δεν είμαστε εξαρτήματα σε ένα μηχάνημα. Είμαστε άνθρωποι, ανθρώπινα όντα, επομένως βρίσκουμε νόημα στις σχέσεις μας με τον πλησίον. Γινόμαστε ολόκληροι, ε, μια ολότητα, όταν συμβάλλουμε σε κάτι που μας υπερβαίνει, σε κάτι που μας ξεπερνά. Οι πολιτικές στο χαρτοφυλάκιό μας ε, υλοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, άρα ώστε να πιο κοντά στους πολίτες και έτσι πρέπει να είναι. Όμως συμφωνώ με όσους από εσάς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκομένους φορείς να αντιμετωπίσουν τις επίγουσες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι. Θέλω λοιπόν να εξυγχρονίσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα από ε, την ε, Πρώην σχολική εκπαίδευση μέχρι τις μεταπτυχιακές σπουδές. Να έχουμε ε, άτομα ε, και δασκάλους ε, με σωστή κατάρτιση, με κίνητρα που να αναγνωρίζεται η αξία τους. Θέλω τα σχολεία, τα πανεπιστήμια να μάθουν τις νέες τεχνολογίες και να υιοθετήσουν νέους τρόπους διδασκαλίας και εκμάθησης και θα πρέπει να εκπληρώσουμε τους στόχους στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020, όλο και περισσότερους ε, αποφύτους ανώτερης ανώτατης εκπαίδευσης, ε, λιγότερη σχολική εγκατάλειψη, γιατί ξέρουμε ότι κάποιος που αφήνει το σχολείο και δεν έχει δεξιότητες ε, θα έχει σημαντικότερα κοινωνικά μειονεκτήματα από τους υπολείπους. Ποιε είναι οι πρώτε μου προτεραιότητε για την επόμενη πενταετία. Πρώτον, πρέπει η εκπαίδευση να μπει στο επίκεντρο των σχεδίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάπτυξη και θέσει εργασία. και ο Ζαν Κλοντ μου ζήτησε να στηρίξω τη δέσμη επενδυτικών μέτρων που θα παρουσιάσει εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του σήμερα. Δεσμεύομαι ενώπιον σας ότι θα ε, συνεχίσω και εγώ και θα, ε, αυτές τις προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου αυτού όχι μόνο τώρα στην αρχή της εντολής, αλλά κάθε χρόνο, όταν δηλαδή θα κάνει τις προτάσεις της, τις συστάσεις αναχώρα προς τα κράτη-μέλη κομισιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να επενδύσουν στους δασκάλους, στις νέες τεχνολογίες, στις νέες διδασκαλίες να εξυγχρονίσουν τις διδακτικές μεθόδους και την διδακτέα ύλη. Ακόμη και όταν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διορθώσουν τα δημόσια οικονομικά τους, είναι ζωτική σημασία να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους στην παιδεία και την κατάρτιση. Δεύτερον, θέλω να εξασφαλίσω ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες θα μπορέσουν να ανθίσουν στον ψηφιακό κόσμο. Η Ευρώπη έχει ηγετική θέση στο δημιουργικό περιεχόμενο και είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει περήφανο. Σήμερα δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι καμία εμπορική διαπραγμάτευση οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα υπονομεύσει το ρόλο της παιδείας και τη μεγάλη σημασία της δημόσιας ενίσχυσης. Θα ήθελα να σας αναφέρω τα λόγια του Jean-Claude Juncker. Δεν θα θυσιάσουμε την πολιτιστική ποικιλομορφία, πολυμορφία της Ευρώπης στο βωμό του ελεύθερου εμπορίου. Και εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του καθεστώτος περί δικαιωμάτων δημιουργού θα προωθήσει και τους καλλιτέχνες μας, του δημιουργούς μας, αλλά και την πολιτιστική πολυμορφία που είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής Ταυτότητα. Όλες οι ευρωπαϊκές δράσεις θα σέβονται την ε, μοναδική φύση της παιδείας μας. Αυτό το ζητάει και η συνθήκη. Τρίτον, θέλω τα πανεπιστήμια μας να γίνουν τα καλύτερα στον κόσμο. Πρόκειται από ιδιαίτερα πολύτιμα ιδρύματα για την Ευρώπη, καθότι είναι πυλώνες της κοινωνίας μας και ζωτική πηγή καινοτομία. Στην Κεντρική Ευρώπη, πριν το 1989, ήταν οχυρά ελευθερίας, κρατούσαν ζωντανή την ελεύθερη σκέψη. Σήμερα πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια πρέπει να ανοίξουν τις θύρες τους στον έξω κόσμο και να προσαρμοστούν στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να βοηθήσει να εξυγχρονιστούν τα πανεπιστήμια μας και να οικοδομηθεί μια νέα σχέση αυτών με την ευρύτερη κοινωνία. Θέλω το τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή παιδεία, έρευνα και επιχειρήσεις, να γίνει μια πραγματική εταιρική σχέση. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα καινοτομία και τεχνολογία, το ΕΙΤ και στις δράσεις μας Μαρίς Σκλοντόσφκα Κιουρί. Το ΕΙΤ είναι ήδη ένα ρηξικέλευθο πρόγραμμα που ήδη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την καινοτομία και είμαι ευγνώμων προ το Κοινοβούλιο που το στηρίζει αυτό το Ίδρυμα, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο για να γίνει μια μεγαλύτερη επιτυχία και οι δραστηριότητέ του να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα το βάλω στο επίκεντρο τη χάραξη πολιτική ε, στην Ευρώπη, γιατί μια καλή πολιτική χρειάζεται σωστή έρευνα, χρειάζεται ενδείξει, στοιχεία. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα ε, υπηρετεί όλους τους τομείς πολιτικής. Ε, είναι πραγματικά το μυαλό ε, στο κέντρο της σκέψης μας και θέλω όλοι να μπορέσουμε να αποφεληθούμε από αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, τέταρτη μου προτεραιότητα. Θα συνεργαστώ στενά με την συνάδελφό μου Μαριάν Τίσεν, Επίτροπο για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, ώστε από κοινού να κάνουμε πάντο δυνατόν για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μόνο τμήμα της λύσης. Πολύ σκληρή δουλειά πρέπει να γίνει και από τα κράτη-μέλη. Όμως ε, θα στηρίξω στεναρά όσες προσπάθειες ε, γίνουν ε, για τη στόχευση, των, στοχεύοντας μάλλον με τους πόρους μου ακριβώς την επίτευξη αυτής, αυτού του σκοπού. Και πιστεύω ότι από κοινού μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Με τη δική σας στήριξη και συνεργαζόμενοι με τα κράτη-μέλη μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να κάνουν τη μετάβαση προς το χώρο εργασίας. Και αυτό το που θα το πετύχουμε με εξυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και συστημάτων κατάρτισης για να μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσει τη αγορά εργασία του 20. Θα στηρίξουμε επίση την ε, εγγύηση για την νεολαία. Ε, θα χρηματοδοτήσουμε νέε εταιρικέ σχέσει μεταξύ πανεπιστημίων, ε, παιδευτικών σχολών, επιχειρήσεων. Θα βελτιώσουμε την ποιότητα των περιόδων άσκηση και μαθητεία και θα δώσουμε στου νέου ανθρώπου όλα τα ωφέλη και τη άτυπη μάθηση. Εκτό αίθουσα δηλαδή. Πέμπτη μου προτεραιότητα θέλω να φέρω και την νεολαία της Ευρώπης ε, ε, μέσα στον κόσμο της χάραξης πολιτικής. Η νεολαία ε, στην Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις άνευ προηγουμένου. Η οικονομική κρίση και έχει οδηγήσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την ανεργία σε πολλές χώρες. Έχει επίσης ε, δημιουργήσει και σημαντικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τη θέση των νέων ε, στην κοινωνία. Οι πολλοί νέοι σήμερα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, συνδεδεμένοι επίσης θα έλεγα σε σχέση με προηγούμενες γενιές χάρη στα νέα κοινωνικά μέσα, αλλά δεν θέλουν πολλές φορές να αρθρώσουν ισχυρό πολιτικό λόγο για την διαμόρφωση της αυριανής κοινωνίας και αυτό θέλω να το αλλάξω. Ο διαρθρωμένος μας διάλογος με την νεολαία έχει αποδείξει την αξία του, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, φτάσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε επαφή και με λιγότερο ε, ευνοημένους ε, νέους. Θέλω λοιπόν να αναπτύξουμε νέες πλατφόρμες για να φτάσουμε σε ένα εκατομμύριο νέους ανθρώπους την επόμενη πενταετία. Αυτό θα σηματοδοτήσει μια πραγματική αλλαγή, στη συμμετοχική δημοκρατία και μια πραγματική στήριξη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να φτάσει τους νέους. Έκτη μου προτεραιότητα θέλω να ε, δώσω μια νέα ε, ανανεωμένη έννοια ε, στον όρο Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Δεν είναι λέξεις αυτές οι δύο, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, λέξη μια συνθήκη. Είναι κάτι παραπάνω από ένα κοινό διαβατήριο, η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Είναι κάτι περισσότερο από το συμπλήρωμα της εθνικής υπηκότητας. Θέλω η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια να είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το ζήσει, να το ανασάνει κατά κάποιο τρόπο. Κάτι το οποίο μας εμπλουτίζει την καθημερινή ζωή, κάτι που βοηθά να οικοδομήσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία θα μπορεί ε, να ε, συνάδει με όλες τις άλλες ε, μορφές και όλες τις άλλες πτυχές ε, της προσωπικότητάς μας. Το χαρτοφυλάκιό ε, μας είναι η καλύτερη δυνατή αφετηρία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός, όλα μας τα προγράμματα, όλες μας οι πολιτικές δημιουργούν την αίσθηση της ηθαγένειας, του ανήκειν. Η ε, Ευρώπη για τους πολίτες, το πρόγραμμά μας θα δώσει συνειδητοποίηση για την κοινή ιστορία, τις κοινέ αξίες, θα κάνει τον κόσμο να καταλάβει τι κάνει για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις λέξεις αθλητισμός, πολυγλωσία δεν θα τις βρείτε βέβαια στο τίτλο του χαρτοφυλακίου ανήκουν στο χαρτοφυλάκι, ανήκουν στα καθήκοντά μου και είμαι υπερήφανο που έχω ευθύνη για αυτά τα δύο ζητήματα. Για πρώτη φορά στον κοινοτικό προπολογισμό ο ευρωπαϊκός αθλητισμός για όλους έχει πλέον 300 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή του για να προστατεύσει τα δικαιώματα των νεαρών αθλητών και παιδιών, για να καταπολεμήσει τη βία, τις διακρίσεις, το ντόπινγκ και τα στημένα παιχνίδια. Θέλω να βοηθήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας να δημιουργήσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και μπορείτε να βασίζεστε στην πλήρη μου υποστήριξη όταν θα δρομολογήσουμε του χρόνου την πρώτη τέτοια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Επίσης θέλω να σας πω και είμαι περήφανος γι' αυτό έχουμε ισχυρά εργαλεία για να προωθήσουμε την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία. Έχουμε το Erasmus Plus, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ένας από τους βασικούς έξι στόχους που έχει είναι η εκμάθηση γλωσσών, η γλωσσική πολυμορφία. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να αξιοποιήσουμε πλήρως τη μεγάλη αυτή ευκαιρία που έχουμε για να προωθήσουμε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης ανεξαρτήτως του αριθμού ε, των ανθρώπων που τις μιλούν. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας καλεί να σεβαστούμε τη γλωσσική μας ε, πολυμορφία και θα συνεργαστώ στενά με τον κύριο Τίμερμαν, ώστε πραγματικά να δικαιώσουμε τις φιλοδοξίες αυτού του χάρτη. Αξιότιμοι βουλευτές, έχω μπροστά μου πολύ σημαντικές προ και για να ανταποκριθώ σε αυτές θα χρειαστώ τη δική σας υποστήριξη. Ακόμη και αν επιτύχουμε, δεν θα δούμε σήμερα όλα τα ωφέλη. Όπως οι αρχιτέκτε των μεσαιωνικών καθεδρικών ναών, μπορεί ίσω να μην ε, ζήσουμε για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα της δουλειά μας. Όμως είμαι έτοιμο για αυτό το χρέο που έχω να επιτελέσω και με, ελπίζω να έλθατε κι εσεί μαζί μου σε αυτό το, το μονοπάτι. Ε, έτσι με μια νότα πιο αισιόδοξη. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να ενθαρρυνθούμε και να αντλήσουμε δύναμη από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Το Εράσμου είναι ε, εμβληματική εφεύρεση Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβολίζει σημαντικέ αξίε τη Ευρώπη, το ανοιχτό πνεύμα, την κινητικότητα, την επιθυμία να συναντηθούμε, να κατανοήσουμε τον πλησίον μα. Οποιοδήποτε άλλο, ε, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πράγμα, πρόγραμμα μα βοηθάει το ε, να χτίσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, κάτι που χρειάζεται η Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα φροντίσω και εγώ να τύχει της χρηματοδότησης που του πρέπει, ε, γιατί γνωρίζετε και εσείς και εγώ ότι ε, δεν είμαστε εμείς ε, οι δύο δηλαδή θεσμοί, τα δύο θεσμικά όργανα που διακινδυνεύουμε τη χρηματοδότησή του. Πρέπει λοιπόν, ε, γιατί ξεκινήσαμε νωρίτερα και το νέο πρόγραμμα, να φροντίσουμε ότι θα φέρει αποτελέσματα για τα 4 εκατομμύρια ανθρώπων που θα σπουδάσουν, θα εργαστούν ή θα δηλώσουν εθελοντέ σε μια ξένη χώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτέ είναι οι προτεραιότητέ με τα επόμενα πέντε χρόνια. Έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε την άκρη να ακούσουμε του πολίτε. Θα είναι τιμή μου να εργαστώ για την ευρωπαϊκή υπόθεση, να υπηρετήσω την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Επίτροπο, ο Επίτροπο, ο δικό σα. Α αρχίσουμε τη δουλειά σα. Ευχαριστώ.